Άρχεται η συνεδρίαση που διακόπηκε στις 18 Σεπτεμβρίου. Κυρίες και κύριοι, δεδομένης της κατάστασης στη Βόρεια Ιρλανδία, ζήτησα από την διάσκεψη των Προέδρων να ζητήσουμε να αποφευχθούν οι επικίνδυνες προκλήσεις και από τις δύο πλευρές και πρέπει να γίνουν προσπάθειες αμέσως για να συνεχιστεί η ειρηνευτική διαδικασία. Και βεβαίως θα πρέπει να εξευρεθεί μια ειρηνική λύση μέσω του διαλόγου. Ζητάμε όμως ε, από όλα τα μέρη να λάβουν μέρος στις ε, νέες διαπραγματεύσεις που ξεκίνησαν στις 16 Οκτωβρίου. Η διαδικασία ειρηνευτική στη Βόρεια Ιρλανδία είναι μια ευρωπαϊκή επιτυχία την οποία θα συνεχίσουμε να στηρίζουμε και το Ευρωπαϊκό Κοινοβούλιο παραμένει τίμιος, ειλικρινής και ανεξάρτητος διαμεσολαβητής και θέλουμε η διαδικασία αυτή να συνεχιστεί επιτυχώς και να στηρίξουμε τη Βόρεια Ιρλανδία να αναπτύξει σταθερούς θεσμούς και οικονομία έτσι ώστε όλοι αυτοί οι άνθρωποι σε αυτό το τμήμα της υπήρους μας να έχουν ένα σίγουρο μέλλον. Κυρίες και κύριοι, θα ήθελα να σας ενημερώσω πως την ε, προηγούμενη πέμπτη η βουλευτής Εβίτα Γκριγκούλ με ενημέρωσε πως ε, εγκαταλείπει την ομάδα του EFDD. Την ίδια ημέρα ενημέρωσε την διάσκεψη των ε, Προέδρων πως πλέον το